beinahe nicht nötig zu erwähnen, aber ohne die Herren links und rechts und da. Και θέλω να πω ότι χωρί τι κυρίε και του κυρίου αριστερά και δεξιά από μένα δεν θα μπορούσα να είχα ε, καταφέρει τόσο καλά να ασκήσω το αξίωμα. Περνάμε όμω χωρί καθυστέρηση στην τη κυρία Παστό για το πρόγραμμα Δάφνη. Τέσσερα λεπτά εισηγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόγραμμα Δάφνη είναι το μόνο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην προστασία των παιδιών, των εφήβων και των γυναικών κατά όλων των μορφών της βίας. Άρχισε το 1997 και αυτό το πρόγραμμα σημείωσε ουσιαστική επιτυχία για όλους τους πληγέντες και καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν. Βλέπουμε λοιπόν τα αποτελέσματα καθώς και τις μελλοντικέ προοπτικές για το πρόγραμμα Δάφνη. Εγκρίθηκε η έκθεση στην Επιτροπή των Γυναικών σχεδόν με ομοφωνία, με μία αποχή δηλαδή. Η συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδες εισηγητές για την ιδιαίτερα θετική συμβολή τους για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Η καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, των εφήβων και των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα και δυστυχώς έχει ακόμη νόημα. Παρατηρούνται νέες μορφές βίας, ε, πρόσφατες μορφές βίας με αυξημένη χρήση των κοινωνικών επιγραμμικών δικτύων καθώς και η βία μέσα στους βρεφονιπιακούς ε, σταθμούς, ε, η κακοποίηση ηλικιωμένων και οι σεξουαλικές επιθέσεις ανάμεσα σε εφήβους. Με την τωρινή οικονομική κρίση και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς Πρέπει να μειώσουμε και το κόστος που συνεπάγονται αυτές οι εγκληματικές ε, πράξεις για το σύστημα υγείας και για το δικαστικά σύστημα. 16 ε, δις το χρόνο. Αυτό είναι το κόστος των εγκληματικών αυτών πράξεων ε, και συμπεριλαμβάνω και την άμεση περίθαλψη, τη δράση των αστυνομικών δυνάμεων, το κοινωνικό κόστος και το οικονομικό κόστος. Πέρσι τον Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Επιτροπή ότι από το 2014 θα ενταχθεί το πρόγραμμα Δάφνη στο γενικότερο πρόγραμμα ε, προστασία ε, των πολιτών, πολιτικής προστασίας. Θα θέλαμε όμως ε, να διατηρήσει το πρόγραμμα την αυτονομία του και θα ήθελα να τονίσω τρία στοιχεία συγκεκριμένα. Πρώτον, να διατηρήσουμε τα θετικά και τα κονδύλια ε, του προγράμματος για την περίοδο 2014-2020 να μην μειωθεί η χρηματοδότηση των προγραμμάτων σε σχέση με το παρελθόν και να εξασφαλιστεί η διαφάνειά του όταν θα ενταχθεί στο μελλοντικό πρόγραμμα για τα δικαιώματα των πολιτών ε, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Ε, οι δικαιούχοι, ε, οι κυβερνητικοί φορείς και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να συνεχίσουν να ενημερώνονται σωστά για τα μέσα χρηματοδότησης και για τους όρους πρόσβασης στο πρόγραμμα. Οι οργανώσεις ε, που είναι κοντά στους πολίτες για πολλά φαινόμενα βίας, δυστυχώς έχουν διοικητικές δυσκολίες. Παρόλα αυτά θα πρέπει να συμμετάσχουν διότι ο ρόλος που διαδραματίζουν είναι θεμελιώδης για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Εξάλλου έχουν και ρηξικέλευθο τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προγραμμάτων. Επίσης χρειάζεται καλύτερος επιμερισμός των προγραμμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη αφετέρου η ε, τακτική συλλογή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για τα διάφορα είδη βία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κέρια σημασία για να έχουμε ε, μια πραγματική εικόνα για τη διάσταση του προβλήματο και να βρούμε τι κατάλληλε λύσει. Τέλο, θα τονίσω το σημαντικό ε, ρόλο τη δράση ευαισθητοποίηση των πολιτών στον τομέα τη υγεία, τη παιδεία, των αστυνομικών δυνάμεων και του δικαστικού συστήματο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Νικολέ έχει μία μπλε κάρτα για σας. Δέχεστε το ερώτημα. Bitte, Frau Nicolai. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felic. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ ε, τον ε, εισηγητή και θα ήθελα να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να βοηθήσει το σχετικό τη σχετική προσπάθεια για αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να προχωρήσουμε μετά το 2014 πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο έχει χρονίσει έχει χρονίσει και ξαπλώνεται για λάβετε υπόψη το κόστος το, ιδίως το κοινωνικό κόστος το οποίο ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και αποτιμήσει πρόκειται για ένα κίνδυνο για την ευρωπαϊκή κοινωνία δεν ήταν ερώτηση αυτό και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι προβλέπονται μόνο ερωτήσεις ε, προς το, τον αγορητή και όχι δηλώσεις. Περνάμε στο Καρδιά. Η Σάλφα Πασέσκο έχει το λόγο πρώτη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω ε, τον συνάδελφο ε, την συνάδελφο συγγνώμη Μπάστος πρόκειται ε, για τον ορθό τρόπο να προσπαθεί κανείς να βρει τον τρόπο να καταπολεμήσει τέτοιου είδους ε, βία. Βία ε, που γίνεται κατοίκων ή αλλού. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την παράγραφο που γράφει το ψήφισμα εκεί στο σήμα τάφη, στο ΖΙΤΑ, ότι η οικονομική κρίση κάνει τα πράγματα χειρότερα για τι ε, γυναίκε. Έχουμε σχετικό πρόγραμμα στη χώρα μου. Ε, ε, τρέχει το Δάφνη 3, έχουμε συγχρηματοδότηση Αυστρία, Τσεχία, Ελλάδα, Σλοβενία. Είναι μια κοινή προσπάθεια. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά μετανάστριε θύματα βία. Με αυτή την πρωτοβουλία εντάσσονται καλύτερα στην κοινωνία, στην ρουμανική κοινωνία και αποτελούν ακόμη και πρωτοβουλία χωρολογή στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Η συνάδελφος Γκυγιώμη έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την κυρία Βαστό για την έκθεσή τη, η οποία νομίζω ότι είναι πολύ πλήρη και αναφέρεται σε όλα τα θέματα που αναφέρθηκαν στην ε, διάμεση έκθεση αξιολόγηση τη Κομισιόν. Η έκθεση αυτή τονίζει το θέμα τη εφαρμογή μέσω των μη κυβερνικών οργανώσεων δομών, μικρών δομών, διαχείριση, ούτω ώστε να τηρηθούν οι στόχοι του προγράμματο. Λυπούμε που δεν υπάρχει πραγματική συζήτηση σήμερα για το θέμα αυτό που θα μας επέτρεπε να ξανατονίσουμε το θέμα της ε, πανταχού παρουσίας της ε, βίας κατά γυναικών νέων και παιδιών. Ιδίω μια που έχουν εντύπωση ότι υπάρχει μια βούληση διαγραφής κάποιων αναφορών στην πορνεία και στην ε, σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα πράγματα που θα πρέπει να διακανονιστούν και δεν είναι ακόμα σαφή. Για να μιλήσουμε για το πώς αναφέρει όλα τα στερεότυπα, θα ήθελα, στερεότυπα, θα ήθελα να πω το θέμα της πρεκοδότησης του προγράμματος αυτού και δεύτερον ότι θέλω να μπορέσει αυτό το πρόγραμμα να καρποφορεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ε, Σας ευχαριστώ. όντω. αυτή η κρίση δεν είναι αποτελεί πρόφαση, ούτως ώστε να μην κάνουμε μια προσπάθεια να λύσουμε αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη. Αντιθέτω, είναι όλο ένα και πιο ξεκάθαρο ότι ε, η κρίση πρέπει να μας οδηγήσει σε περισσότερες προσπάθειες. Άρα θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθεια και για να αντιμετωπίσουμε την βία των γυναικών και για μένα αυτό είναι βασικό θέμα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσει το κοινοβούλιο μας. Είναι και θέμα οικονομικού κόστος, όμως από την άλλη μεριά είναι αλήθεια ότι η βία ε, προκαλεί ακόμα και οικονομικές δυσμενείς συνέπειε. αλλά πέραν αυτών των συνεπειών θα πρέπει να δούμε ε, το θέμα της ουσία ακριβώς όπως το είπε η συνάδελφος. Δεν είναι δυνατόν αυτή η συζήτηση να μας οδηγεί σε ιδεολογήματα, ε, να μας οδηγεί σε μια λογική στιγματισμού των γυναικών θυμάτων ε, και θα πρέπει να προσέξουμε να είναι πιο προστατευμένες και όχι πιο ευάλωτες οι γυναίκες και έκθετες στην απειλή της βίας. Επομένως ε, θα πρέπει πέραν όλων των άλλων θεμάτων να μην ξεχνούμε την ουσία του θέματος, δηλαδή την δυσμενή διάκριση που αφήσατε σε πάρα πολλούς χώρους της κοινωνίας, το μη κοινωνίας και Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ του επόμενου ομιλητέ να τηρήσουν τον χρόνο χωρί που έχουν, α, γιατί αλλιώ έχουμε τεράστια καθυστέρηση. Συνάδελφο Σούσκοβα έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω το περιεχόμενο της έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα Δάφνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σημειωθεί πρόοδος ε, για το τόσο επιτυχημένο και σημαντικό πρόγραμμα, διότι συνιστά και την ε, ε, βασική δύναμη κρούση που έχουμε για την προστασία των γυναικών, των εφήβων και των παιδιών. Πρέπει να εξασφαλίζουμε προστασία για τα θύματα οικογενειακής και άλλων μορφών Τα θύματα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση Στι κατάλληλε επιδοτήσει και στα κέντρα υποδοχής. Ε, Διαπιστώνατε σε πολλά μέρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Πιστεύω ότι χάρη στο πρόγραμμα Δάφνη θα έχουμε και άλλα πολλά ε, επιτυχημένα υποπρογράμματα. Εγώ συμφωνώ με διάφορε δράσει που προτείνονται, παραδείγματο χάρη ίσω επιμερισμό, δίκαιος μάλλον επιμερισμό των προγραμμάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λιγότερη γραφειοκρατία, απλό απλοποίηση της διαδικασίας ε, υποβολής αίτησης ε, για χρηματοδότηση και βοήθεια προς τις μικρές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Ζαπόρσκα έχει το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ κυρία Μπαστός για την έκθεση αυτή όταν εξετάζουμε το θέμα των πρωτοτήτων για το μέλλον αξίζει να εξετάσουμε το παρελθόν και να επιθυμίσουμε τις ε, ε, πρωτοβουλίες που οδηγούν σε αποτελέσματα. Μεταξύ αυτών είναι και το πρόγραμμα Δάφνη. Το πρόγραμμα Δάφνη είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πολλά μπορούν να επιτευχθούν ε, όταν βρίσκεται εκτός της εμβέλειας άλλων οργάνων. Πρόκειται για το θέμα των γυναικών, των παιδιών που υπόκειται σε βία και δεν πρόκειται μόνο για φυσική βία αλλά και απειλές, ψυχολογική βία, παρενοχλήσεις κλπ. κλπ. Αυτά όλα ε, αποβαίνουν σε βάρος της ψυχολογικής κατάστασης των λογοτομων και ε, το πρόγραμμα Δάφνη μπορεί να αντιμετωπίσει και αυτά τα προγράμματα και επίσης ε, τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων στο διαδίκτυο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Επόμενος και τελευταίος ομιλητής. Γιατί προσπαθούμε να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των φίλων. Ο κύριος Πρέντεργκας. Α, όχι, η κυρία. Η κυρία Πρέντεργκας. συγγνώμη. I shouldn't apologize about my gender. Ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να ζητάω συγγνώμη για το φίλο μου. Ε, είναι σημαντικό το πρόγραμμα Δάφνη να ε, ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα ηθαγένειας ε, και να εστιάσουμε την προσοχή μας στις μελλοντικές ε, πρωτοβουλίες όπως είχαμε προσπαθήσει και σε προηγούμενα προγράμματα, Δάφνη. Πρέπει να εστιάσουμε τη δράση μα ε, στι μη κερδοσκοπικέ οργανώσει και τι μικρέ μη κυβερνητικέ οργανώσει που είναι σημαντικέ για να επιτύχουμε του στόχου μα. Στη δική μου τη χώρα, διάφοροι φορεί έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα Δάφνη και σχετικέ ε, πρωτοβουλίε που χρηματοδοτούνται μέσα από το Δάφνη για την προστασία των γυναικών, των εφήβων και των παιδιών. Ναι. Πρόκειται για την πρωτοβουλία αξιοπρέπεια ε, όπου υπήρχε συνεργασία μεταξύ διαφόρων κοινωνικών εταιρεών για να βελτιωθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες ε, υπέρ των θυμάτων ε, της σεξουαλικής κακοποίησης, ώστε να έχουμε και μια γραμμή βοήθειας για αυτά τα παιδιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τη δράση αυτών των φορέων, φορέων συγγνώμη, και παρεμφερών φορέων που δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην Επιτροπή κυρία Γεωργίευα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, την κυρία Μπάστος και τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών, διότι συνέταξαν μια ιδιαίτερα ισορροπημένη έκθεση. Σε ευχαριστώ για τη διαρκή υποστήριξή τους προς τα προγράμματα Δάφνη. Βάσει του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να καλύψει όλες τις δράσεις που υποστηρίζονται και υλοποιούνται τώρα μέσα από το πρόγραμμα Δάφνη, να τα εντάξει λοιπόν στο ε, πρόγραμμα Ιθαγένειας και Δικαιωμάτων των Πολιτών. Να απαντήσω τώρα σε ερωτήσεις. Υπό το νέο πρόγραμμα όλες οι στόχοι, όλες οι δράσεις που υπάρχουν στο πρόγραμμα Δάφνη θα υποστηριχθούν και τα κονδύλια σε αυτό τον προϋπολογισμό, στο νέο προϋπολογισμό, είναι απολύτως αντίστοιχα προς στα κονδύλια του προηγούμενου πλαισίου. Βάσει λοιπόν του πολυετούς πλαισίου επικεντρωνόμαστε στην απλούσταση, στην ευελιξία και στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Στοχεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη των βέλτιστων δυνατών συνεργειών ανάμεσα σε τρεις δραστηριότητε. Καταπολέμηση τη βία, προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Αυτό το πρόγραμμα θα καλύψει τις αναδυόμενες νέες μεγάλες προκλήσεις ε, που αναφέρονται μερικώς μέσα στην έκθεση της κυρίας Μπάστο. Θα ήθελα να τονίσω ότι το νέο πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό σε όλες τις ε, νομικές οντότητες, σε όλα τα κράτη-μέλη, για όλες τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που έχουν διενεργηθεί και χρηματοδοτηθεί βάσει του προγράμματος Δάφνη 3. Το νέο πρόγραμμα θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τη δράση ως προς τη διαχείριση των προβλημάτων και να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και να αντιμετωπίσει τις ατέλειες ε, που διαπιστώθηκαν στην ενδιάμεση έκθεση αξιολόγηση ε, του Δάφνη 3 και που αναφέρονται μέσα στην έκθεση. Παραδείγματο χάρη, καλύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων. Ε, Επίση, ε, γεωγραφική κατανομή των προγραμμάτων. Οι δικαιούχοι, οι άμεσοι δικαιούχοι θα υποφεληθούν από την αναβαθμισμένη διαχείριση των προγραμμάτων. Θα είναι ταχύτερε, λιγότερο γραφειοκρατικέ, πιο ομοιόμορφε, ευκολότερε οι διαδικασίε για να επιτύχουν τη χρηματοδότηση. Το 2012 Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναβαθμίσει ρυθμίσει και το ΚΙΤ Δάφνη 2012, διάφορα εργαλεία δηλαδή για την καταπολέμηση τη βία, θα μα βοηθήσει ούτως ώστε να διαδίδουμε τα αποτελέσματα των προγραμμάτων που έχουν αναλάβει οι εθνικοί και περιφερειακοί φορεί, ώστε στα πλαίσια του νέου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα ω πρότυπο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων προγραμμάτων και σε άλλου τομεί. Θα ήθελα να τονίζω επίση ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια ότι προφανώ ε, Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε άλλε χώρε για την καταπολέμηση των ε, ε, αξιόπινων πράξεων κατά των γυναικών αν δεν έχουμε τακτοποιήσει τα ε, δικά μας προβλήματα και θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την εισηγήτρια και επιστρέφω τώρα τα δύο λεπτά που σας είχα κλέψει από την προηγούμενη παρέμβαση. Ευχαριστώ. Θαυμάσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνω τη συζήτηση του έμενος αυτό σημείο της διάταξης και περνάμε στο επόμενο σημείο την έκθεση Νικολάη σχετικά με τη θέση των γυναικών στους πολέμους. Και θα ήθελα να δώσω την εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι.